Ε, τις εσωτερικές συγκρούσεις της Ουκρανίας. Ε, α εκπληρώσουμε εμεί τα καθήκοντά μα και θα ανταμυφθούμε από, το, από τις ίδιες μελλοντικές εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Σεβερίν από πλευρά των φιλελευθέρων. Ε, κυρία Βαλέαν. Yes, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε.